Ευχαριστώ. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, Πρόεδρων Επιτροπών, μέλη του Κοινοβουλίου, ευχαριστώ για τις ερώτησεις σας. Στις τελευταίες εβδομάδες συνάντησα όλες τις πολιτικές ομάδες και τους πολιτικούς, τους συντονιστές των ομάδων που μπόρεσα, ώστε να επικεντρωθούμε στα πραγματικά θέματα που αναφέρθηκαν κατά διάρκεια αυτής της, ακρόαση. ακρόασης. Ο ψηφιακός τομέας έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στην πρόθεση της ανάκαψης στη δημιουργία θέσεων εργασίας και των επενδύσεων στην Ευρώπη. Ο ψηφιακός κόσμος είναι παντού. Προοδεύει, προχωράει κάθε μέρα και η Ευρώπη ακριβώς θα πρέπει να τον ακολουθήσει. Αν με αποδεχτείτε ως αντιπρόεδρο η ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς για την Ευρώπη θα αποτελέσει την κύρια προτεραιότητά μου, όπως ακριβώς αναφέρεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε ο υποψήφιος πρόεδρος της Κομισιόν κ. Γιούνκερ, ώστε όχι μόνο να ενισχύσουμε την ε, οικονομία μας, αλλά και για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, αλλά και για να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των πολιτών μας και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προωθήσουμε το ψηφιακό περιβάλλον στην Ευρώπη, θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε την ε, ανασφάλεια Δικαίων και θα πρέπει να δημιουργήσουμε ίσες ευκαιρίες για όλους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε την ύπαρξη ευθύνη στο ψηφιακό περιβάλλον και να προστατεύσουμε τα ιδιωτικά και τα εμπορικά δεδομένα. Σημαίνει ότι θα πρέπει να αφαιρέσουμε τα αναπομείναντα εμπόδια που αφορούν σήμερα τον κατακαιρματισμό της ψηφιακής αγοράς. Νομίζω ότι η νέα ψηφιακή αγορά είναι αυτό που επιθυμούν πραγματικά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Υψηλές ταχύτητες, συνδέσεις για όλους, απάλληψη φραγμών διασυνοριακών, όλα αυτά μέσω συνδεδεμένων και σύγχρονων υποδομών. Για να ανταπακριθούμε λοιπόν στις προσδοκίες και στα αιτήματα, στις απαιτήσει των πολιτών των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτίθεμαι να εργαστώ όσο πιο διαφανώς γίνεται με διαβουλεύσεις, με μέσω εταιρική και σε ένα πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης μαζί σας. Θα διατηρήσω ένα συνεχώ, συνεχή και τακτικό διάλογο με όλες τις επιτροπές. Ευχαριστώ πολύ. Υποψήφια Επίτροπε, σας ευχαριστώ εκ νέου για μια τόσο μακρά ακρόαση δεν ήσασταν και πολύ καλά τις τελευταίες εβδομάδες. Ε, καλύψατε τεράστιο φάσμα θεμάτων, Από όταν ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής και ανέλαβαμε την ευθύνη για την ψηφιακή νέα αγορά, ήταν σαφές ότι συνάδελφοι όχι αυτής της Επιτροπής, αλλά από όλο το Κοινοβούλιο, θεωρούν ότι ο ψηφιακός κόσμος είναι ένας χώρος που δεν ζει κάπου ξεχωριστά, αλλά είναι ένας χώρος όπου κινείται η οικονομία μας και εκεί πρέπει να αναπτυχθεί και να οικοδομηθεί και είναι κάτι που επηρεάζει κάθε τι που κάνουμε και θα κάνουμε στο μέλλον. Και είμαστε έτοιμοι να προσπαθήσουμε να στερνιστούμε τις διάφορες αυτές προκλήσεις και πραγματικά να κερδίσουμε τα ωφέλη από μια ασφαλή αλλά ζωντανή ψηφιακή αγορά, ψηφιακό κόσμο. Προσβλέπουμε αύριο στην αξιολόγησή σας δεν χρειάζεται να κάνετε δημόσια κρόαση πριν κάνουμε εμείς την αξιολόγησή μας. Η δημόσια κρόαση διεξήχθη εδώ. Αν θέλετε να κάνετε κάποια επικοινωνία, έχει επικοινωνία στο διαδίκτυο, καλώς, αλλά η αξιολόγηση θα βασιστεί σε αυτή την ακρόαση και όχι σε μελλοντικές συζητήσεις στο διαδίκτυο. Έληξε το τρίωρο και οι τρεις εμπλεκόμενες επιτροπές θα συναντηθούν, θα συναντηθούν αύριο το πρωί 11 το πρωί οι συντονιστές. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς θα διεξαγάγει μια συζήτηση στα πλαίσια των συντονιστών μας πριν από αυτό. Αύριο στις 11 στην 6Q2 για να αποφασιστεί δημοκρατικά το πώς θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλό σας βράδυ.